Καλή σα μέρα. Περνάμε στι επεξηγήσει ψήφου των ψηφισμάτων που πριν από λίγο εγκρίναμε. Θα ακούσουμε πρώτα τι επεξηγήσει ψήφου ε, επί τη εκθέσεω Μορέλ για την μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ιορδανία. Παρακαλώ όσοι εγκαταλείψουν την αίθουσα να το κάνουν αθόρυβα για να μπορέσουμε να ακούσουμε τους ομιλητές. Πρώτος ο κύριος Γίζη Πόσπισιλ. Παρακαλώ, σας ακούμε κύριε Πόσπισιλ. Mr. Pospisil, take a floor, please. Παρακαλώ κύριε Πόσπισιλ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.